Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Δεν είναι βέβαια εδώ πολλοί συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μην τιμωρήσουμε όσους φτάνουν στην ώρα τους. Σας καλωσορίζω όλους λοιπόν στην πρώτη συνεδρίαση μετά το μεσημεριά, το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ελπίζω να περάσατε ευχάριστες διακοπές, να μαζέψατε δυνάμεις, γιατί μας περιμένει δύσκολο έργο. Θέλω να καλωσορίσω ένα νέο μέλος στην Επιτροπή μας, δεν είχαμε δείξει στην προηγούμενη συνάντηση βέβαια έχουμε και έναν, αντι, έναν αντικαστάτη της κυρίας Κομοντίνη, τον κύριο Ντίματς. Ελπίζω να ε, πρόφερα σωστά το όνομά σα κύριε Ντίματς, και ελπίζω να έχουμε μια καλή και ευχάριστη συνεργασία. Λοιπόν, έχουμε πρώτα την έγκριση της σημερινής ημέρησιας διάταξης. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Η κυρία Ρεμπέτσκα που θα μιλήσει είναι εξχρονισμό της, πολιτικής, της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μόλις εμφανίστηκε στις Βρυξέλλες, μόλις φτάσει στις Βρυξέλλες και δεν είναι ακόμα εδώ, οπότε θα έλεγα να μιλήσουμε πρώτα ε, για την έκθεση σχετικά με την ομάδα monitoring του Brexit. Ας δούμε αυτό το θέμα λοιπόν πρώτα. Μικρή αλλαγή λοιπόν στην εμείς εκτός αν, δεν, αν έχει κάποιος αντίρρηση. Μάλλον όχι. Οπότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται μέσα σε διάταξη με αυτή τη μικρή αλλαγή. Το δεύτερο σημείο είναι η έγκριση των πρακτικών. Το σχέδιο πρακτικών στις 4 Μαΐου και 24-23 Ιουνίου και 29 Ιουνίου όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο, στα εγγραφά σα. Έχετε σχόλια για τα πρακτικά. Όχι. Οπότε θα πρότεινα να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορείτε ακόμα εντός της ημέρας, εντός της συνεδρίας, της συνεδρία να αναφέρετε κάποιες αντιρρήσεις. Λοιπόν, σημείο 3, ανακοινώσει του Προέδρου. Η γλωσσικό καθεστώς καλύπτει μια σειρά παρόλους να και τα ελληνικά. Μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε ελληνικά σας θυμίζω ότι υπάρχει web streaming σήμερα. Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι και οι αποφάσεις των συντονιστών της 11ης Ιουλίου έχουν σταλεί ήδη σε όλα τα μέλη από τη 12η Ιουλίου και θα θεωρηθούν επισήμως εγκεκριμένα διότι μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία που ήταν ε, προθεσμία μάλλον, 14 Ιουλίου, δεν υποβλήθησαν ενστάσεις. Έχω απευθύνει ήδη χαιρετισμό στα νέα μέλη. Έρχομαι σε μια ανακοίνωση που ίσως ε, σας φανεί λιγότερο ευχάριστη. Θέλω να σας επισημάνω ένα μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για το προπολογισμό του 2018. Το Συμβούλιο προτείνει περικοπή κονδυλίων της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Projecting Europe. 1,5 εκατομμύρια 6 εκατομμυρίων θα εξοικονομηθούν από το υποπρόγραμμα Media και 4,5 εκατομμύρια από το υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Όσον αφορά πάλι τα Media, έχουμε ζητήσει εμείς 13 εκατομμύρια παραπάνω και 14,5 για τα ξεκινώντας από την βάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τα νούμερα αυτά φαίνεται καθαρά ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των θέσεων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ώστε δεν μπορώ παρά να κάνω το σχόλιο ότι έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο δεν αντιλαμβάνεται την σημασία του προγράμματος για το οποίο μιλούμε. Πώς είναι δυνατόν να τους έρθει η ιδέα σε περιόδους όπου ενισχύεται ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός να μειώσουν, να περικόψουν κονδύλια για τέτοια προγράμματα που ενισχύουν κοινέ αξίες σε ένα κοινό χώρο πολιτισμού. Βρίσκω ότι μια τέτοια ιδέα είναι και παράτολμη και ανόητη. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα Media έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, πολύ μεγαλύτερη από τα κονδύλια που προβλέπονταν Εάν θέλουν λοιπόν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την απογοήτευση του κόσμου, α κάνουν αυτό που προτείνει το Συμβούλιο. Όμως, στην βάση της αιτιολόγησης για την περικοπή των κονδυλίων για το πρόγραμμα πολιτισμός, βλέπουν ότι ο προγραμματισμός δεν παίζει για αυτού κανένα ρόλο. Όταν λένε ότι το 2017 δεν απεροφήθησαν όλα τα κονδύλια για χωρί να ρωτήσουν γιατί, θεωρώ ότι η αιτιολόγηση του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ αδύναμη. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα 2017 εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και γι' αυτό δεν μπόρεσε να γίνει εξυπηρέτηση των κονδυλίων. Έρχονται τώρα λοιπόν και απευθύνουν την μομφή ότι δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια. Αυτό, για να το πω καθαρά για μένα, είναι ανέβεια. Η προτινόμενη περικοπή κονδυλίων στο πρόγραμμα πολιτισμός παραβιάζει και τη συμφωνία με το Κοινοβούλιο για, την, για το έτος πολιτιστικής κληρονομίας του 2017. Είχαμε συμφωνήσει να δοθούν 4 εκατομμύρια νοπόχρημα. Τώρα, τα χρήματα που πήραν από το υποπρόγραμμα πολιτισμός και τα ανακτούν μάλιστα τώρα, σύμφωνα με τον δικό τους προγραμματισμό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από εμάς τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Ίσως να διαθέτουμε λοιπόν κονδύλια αρκετά για το έτος πολιτιστικής κληρονομίας, αλλά να προχωρούν τώρα σε περικοπές κονδυλίων θεωρώ ότι είναι απολύτως απαράδεκτο και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε όλοι και όλες μαζί μου. Για το 2016, 11% όλων ε, προσώπων που έβαλαν αιτήσει έλαβαν κάποια ενίσχυση. 89% έμειναν με άδεια χέρια. Και αυτό όχι επειδή δεν ήταν καλά τα προγράμματα ή τα σχέδια που υπέβαλαν, δηλαδή δεν υπήρχαν κονδύλια. Με απλά λόγια έχω να πω στο Συμβούλιο ότι αυτά δεν είναι πράγματα. Και στις παραπέρα διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό σας παρακαλώ όλες και όλους να ενισχύσετε την προσπάθειά μας μέσα από όλες τις πολιτικές ομάδες ώστε σε αυτές οι περικοπέ κονδυλίων να μην γίνουν δεκτέ από το Κοινοβουλίο. Αυτέ δηλαδή που προτείνει το Συμβούλιο. Και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπέρ τη ενίσχυση των κονδυλίων, Όπω έχουμε προτείνει. Ελπίζω ότι θα βοηθήσετε όλοι και όλε με όλε σας τις δυνάμεις, ώστε αυτή η επίθεση εντό εισαγωγικών κατά του πολιτισμού να μην επιτύχει από πλευρά του Συμβουλίου. Καλά λοιπόν, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι παραπέρα διαπραγματεύσεις αλλά για να είμαι ειλικρινής συγκλονίστηκα, σας το λέω καθαρά, όταν άκουσα τα νέα αυτά για το τι σχεδιάζει και προτείνει το Συμβούλιο. Και ήθελα βεβαίω να σας ειδοποιήσω κιόλα ώστε να τα γνωρίζετε. Βεβαίω ορισμένοι μπορεί να τα γνωρίζετε ήδη. Αυτές λοιπόν ήταν οι ανακοινώσει μου ως Προέδρου και νομίζω να προχωρήσουμε αμέσως στο θέμα 4 της ημέρης της διάταξης, δηλαδή την έκθεση για την πρώτη συνάντηση της ομάδας παρατηρητών Brexit στο γεύσκι του Λαϊκού Κόμματος. Όρισαν τα μέλη για την Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευρά της Επιτροπής Πολιτισμού, δηλαδή της πορείας των ε, διαπραγματεύσεων για την Βρετανική έξοδο, ε, για τα τμήματα εκείνα που αφορούν την Επιτροπή Πολιτισμού για το Brexit θα διαβάσετε και εσείς τι εφημερίδες ότι έχουν ήδη γίνει τρεις γύροι διαπραγματεύσεων. Ο τρίτος γύρος έγινε μόλις την προηγουμένη εβδομάδα. Έχουν εκδοθεί και κάποια έγγραφα, δημοσιεύτηκαν μάλιστα κάποια έγγραφα και η monitoring ομάδα του Brexit έκανε την πρώτη συνάντηση λίγο πριν από τις θερινέ διακοπές στο Στρασβούργο. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Στογεύσκη να ενημερώσει την Επιτροπή Πολιτισμού και ίσως να πει και λίγα λόγια σχετικά με τον τρόπο εργασίας της ομάδας παρακολούθησης της ε, Brexit, σε τι δηλαδή έχετε συμφωνήσει και ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά ορόσημα στην εργασία σας. Κύριε Στογεύσκη, σας δίνω το λόγο τώρα για πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εγώ, αλλά θέλω να μιλήσει και... Θέλω να περιμένουμε μάλλον και τον κύριο Κομπάσκα. Αλλά θα είμαι σύντομο. Δυστυχώ ε, δεν έχω και πολλέ καλέ ειδήσει και γι' αυτό αναγκαστικά δεν έχω να πω και πολλά. Η ομάδα εργασία μα που έχει χαρακτήρα ας πούμε παρατηρητού έχει τρεις βασικά αρμοδιότητες και καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια ώστε να παραμείνουμε εντός των ορίων μας, των ορίων των αρμοδιοτήτων μας, δηλαδή να συμβάλλουμε για την διατύπωση του τελικού ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, να μπορούμε να απαντούμε σε ερωτήσεις που προκύπτουν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και η τρίτη μας αρμοδιότητα είναι αυτή της ανάλυσης και συζήτησης των εγγράφων για... που εκδίδονται για τον Brexit και που ε, άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, έγιναν ήδη τρεις γύροι διαπραγματεύσεις, πραγματικότητα δύο, διότι η πρώτη συνάντηση της 9ης έκτου στην ουσία δεν ήταν παρά η έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας και δεν έγινε συζήτηση επί της ουσίας. Στις 17 Εβδόμου και στις 28 επίσης ξαναμιλήσαμε. Στις 17 δεν είχαμε συζητήσει, δεν συζητήσαμε τίποτα που να είχε σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες. Στις 28 όμως Αυγούστου, 8, κάποια σημαντικά θέματα συζητήθηκαν που έχουν ενδιαφέρον δηλαδή και για την Επιτροπή Πολιτισμού. Και έχω να σας πω το εξή Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit κινούνται μέσα σε πολύ θα έλεγα δυσμενείς συνθήκες. Εγώ διαπιστώνω να υπάρχει μια έλλειψη προετοιμασίας. Βλέπω να κυριαρχεί μια διαδικαστική αναρχία. Αυτό δεν ευνοεί την ε, καλή διεξαγωγή των εργασιών, ούτε και να προκύψουν και καλά αποτελέσματα. Από τα θέματα που συζητήθηκαν στον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων, αυτά ήταν κυρίως για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, διπλωμάτων, πτυχίων κλπ. Και μπορώ να πω ότι την τελευταία στιγμή του γύρου αυτού διαπιστώθηκαν ότι τα όσα ισχύουν έως τώρα, όσα δηλαδή αναγνωρίζονται ως τώρα, προσόντα, πτυχία κλπ, θα πρέπει να συνεχίσουν να αναγνωρίζονται. Δηλαδή όσα ήδη έχουν αποκτηθεί πριν από το πέρας των διαπραγματεύσεων για το Brexit και όσα θα έχουν αποκτηθεί δηλαδή μέχρι τότε, αυτά θα αναγνωρίζονται. Ε, πρόκειται για ένα επίτευγμα μικρό βέβαια, αλλά πρέπει να συζητηθεί και το τι θα γίνει με τους σπουδαστέ και μαθητές εκείνους που φοιτούν σε πανεπιστήμια ή σχολεία ήδη και που θα τους πιάσει το Brexit. Το ερώτημα είναι θα αναγνωριστούν τα πτυχία τους ή όχι. Από αυτά που ξέρουμε φαίνεται πως ε, σπουδάζουν πάρα πολλοί νέοι και νέες στη Μεγάλη Βρετανία και όχι το αντίστροφο, δηλαδή δεν είναι πολλοί Βρετανοί φοιτητέ σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να ε, διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας στον τομέα αυτό διότι είναι ένα θέμα το οποίο θίγει την νέα γενναία και επομένως μια ομάδα προσώπων που είναι ευάλωτη. Άρα πρέπει να παραμείνουμε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε λάβει πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα των Βρετανικών Πανεπιστημίων και ποια θα είναι η πορεία τους μετά από την Βρετανική έξοδο, αλλά ακόμα δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση, καμία τελική απόφαση δηλαδή στις διαπραγματεύσεις. Στις 18 Ενάτου θα γίνει ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων και εφόσον λάβω σχετικά έγγραφα θα συγκαλέσω και πάλι την ομάδα μας, ομάδα παρατήρησης και θα συζητήσουμε τις νέες αυτές πληροφορίες που θα προκύψουν, θα τις αναλύσουμε και θα τις ε, συζητήσουμε υπό το φως των εξελίξεων. Τώρα, για τον τρόπο εργασίας. Εγώ προτείνω τα μέλη μας να περιοριστούν αυστηρά στις αρμοδιότητες μας, σε αρμοδιότητες τις δικές μας. Η δική μας λοιπόν ομάδα παρατηρητών αντιμετωπίζει ερωτήματα, θέματα τα οποία είναι νέα. Γίνεται προσπάθεια να μας ε, φορτώσουν και κάποια άλλα θέματα, αλλά μια στιγμή δεν είμαστε ε, ένα είδο κάλαθος αχρήστων όπου καταλήγουν όλα τα άλλα όσα δεν δέχονται να συζητήσουν άλλοι. Εγώ θα προσπαθήσω, θα φροντίσω ώστε η συζήτησή μας να παραμείνει αυστηρά εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων μας. Βεβαίω το όριο, τα όρια αυτών των αρμοδιοτήτων δεν είναι ανάγκη να είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρά. Αλλά εφόσον πρόκειται για παράδειγμα για τις συμβάσεις εργασίας των προσώπων που εργάζονται στον πολιτισμό, ε, εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχολές τεχνών ε, ή προγράμματα όπως το Creative Europe η Ευρώπη για τους πολίτες κλπ. Αυτά ναι. Πέραν των ελευθεριών που αφορούν τους πολίτες διαπιστώνω ότι τα θέματα του πολιτισμού η συζήτησή τους δηλαδή κάπως αναβάλλεται δηλαδή τα δικά μας εντός εισαγωγών θέματα θα συζητηθούν του χρόνου τον Σεπτέμβριο, έτσι ακούσαμε. Τώρα, εμείς θα παρακολουθούμε βέβαια, όπως είπα, όλες τις εξελίξεις. Δεν είναι δυνατόν κάποια σημαντικά θέματα τα οποία ανήκουν στις δικές μας αρμοδιότητες να παραμείνουν εκτό. Τώρα, για τα θέματα, για τα οικονομικά θέματα. Έχω πληροφορίες ότι τα θέματα τα οικονομικά και ιδίω τα δημοσιονομικά θεωρούνται από τη Βρετανική πλευρά πάρα πολύ σημαντικά και πολύ καυτά. Και αυτά βεβαίω έχουν σχέση και με την εκστρατεία που προηγήθηκε λήφθηκαν τότε πολύ σοβαρές και βαριές αποφάσεις. Μιλούν για την συνεισφορά της ε, Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, είχαν μιλήσει, είχαν πει τότε ότι η συνεισφορά αυτή θα αφιερωθεί πλέον για τη βελτίωση των ιατρικών υποδομών. Όμω αυτό κάτι τέτοιο αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατο. Γι' αυτό και θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση και γύρω από τι υποχρεώσει τη Μεγάλη Βρετανία απέναντι στι υπόλοιπε χώρε μέλη τη Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί και στις συζητήσεις και για τις διάφορες εμπορικές συμφωνίες που ναι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αλλά μπορεί ωστόσο να μας ενδιαφέρουν. Μετά τον νέο γύρο, όπως είπα, των διαπραγματεύσεων θα ακολουθήσει νέος γύρος εργασίας της δικής μας ομάδας. Μιλούμε για τα δικαιώματα των ε, σπουδαστών που βρίσκονται τώρα σε βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και βεβαίω και για τα πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν αποκτήσει τα, τα ε, πτυχία αλλά για αυτού βέβαια δεν αμφισβητείται το θέμα. Έχω τώρα και κάτι άλλο σημαντικό για τον προπολογισμό. Βεβαίω και είναι σκάνδαλο η προσπάθεια που γίνεται περικοπής, αφαιρεση δηλαδή, κονδυλίων. Και η κυρία Σίλβια Κώστα έχει συζητήσει θέματα πολιτικής κληρονομίας. τα 4 εκατομμύρια για την υποστήριξη των προγραμμάτων αυτών θα έρχονταν από νοπά χρήματα και τώρα προσπαθούν να τα εξεύρουν μέσα από άλλα στοιχεία του μέσα από άλλα κονδύλια του προπολογισμού. Αυτό όμω είναι αντίθετο με τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρο Κάμερ ευχαριστώ για την τελευταία σα παρατήρηση όσον αφορά τον προπολογισμό. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πράγματι εκτό τη συμφωνία που, που είχαμε κάνει μάλλον με το Συμβούλιο. Και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε και να το ξαναπούμε. Τώρα, εκ των συντονιστών, αν βλέπω καλά είναι μονάχα παρούσα η Σίλβια Κώστα, η οποία λαμβάνει το λόγο για δύο λεπτά και ναι, ο εισηγητή είναι του Λαϊκού Κόμματο, έτσι είναι. Σκιώδη εισηγητής, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε όλοι από τις διακοπές. Ένα-δύο πράγματα που ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστώ τον κύριο Τρολογεύσκη διότι αναφέρθηκε ε, σε αυτή την πρώτη συνάντηση την οποία της οποίας έκανε μια πολύ καλή περίληψη υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι σημαντικά για μας στο έγγραφο αυτό όπου αναφέρεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της αναγνώρισης των πνευματικών προσόντων. Επίσης, με βάση αυτό το έγγραφο αναγνωρίζεται, αναγνωρίζεται και οι δεξιότητες στα προσόντα τυπικών τρίτων χωρών και αυτό είναι πολύ σημαντικό βεβαίως. Πολλά ακόμα παραμένουν ασαφή σε ό,τι αφορά τις αλλά θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην απώλεια της άδεια παραμονής. Εγώ δεν είμαι νομικός Όμω, μίλησα με εμπειρογνώμονες και μου είπαν ότι οι άδειες παραμονές στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι δύσκολο να χορηγηθούν. Δίνεται δηλαδή ε, η άδεια ε, κατοικίας, αλλά όχι άδεια παραμονής. Η άδεια παραμονής χορηγείται μόνο όταν κάποιος έχει ζήσει ήδη πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, έτσι μου είπαν. Θα πρέπει να εξεταστεί. Τώρα, το γεγονό ότι μετά από δύο χρόνια θα χάνεται η άδεια παραμονή και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τι θα γίνει με του διάφορου ερευνητέ, του πανεπιστημιακού, ε, σε αυτού ε, που εργάζονται σε διάφορα project. Θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξουν εξαιρέσει. Ε, διότι είναι κάτι που συνδέεται με την άσκηση του επαγγέλματος, την ελεύθερη άσκηση ενό επαγγελματο, μια επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα, κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να ληφθούν υπόψη ε, αυτοί οι οποίοι ήδη διαμένουν πέντε χρόνια ε, για να μην είναι προσωρινή για αυτούς η άδεια. Εμείς θέλουμε να συμπεριλάβουμε εδώ και τους φοιτητέ που αλλάζουν καθεστώς, δηλαδή που ήταν φοιτητέ και μετά στη συνέχεια γίνονται καθηγητές. θα πρέπει εκεί να γίνεται αυτόματα αυτό. Και κάτι άλλο. Το θέμα των παροχών. Υπάρχουν πολλές παροχές ε, για φοιτητές, ε, ε, ερευνητές, υπάρχουν ε, στεγαστικά επιδόματα κτλ. κτλ. Θα πρέπει να δούμε εκεί τι εμπίπτει στη δική μας τα και τι όχι. Τώρα για τον προπολογισμό ούτως ή άλλως Αύριο θα γίνει μια συνάντηση με τους συντονιστές για το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους της ε, Πορτικής Κληρονομιάς και εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το θέσουμε το θέμα από πλευράς Κοινοβουλίου διότι δεν αιτιολογεί της καμία περίπτωση αυτή η περικοπή η οποία είναι στα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Ε, Σαμπίνε όχι δεν θέλει να μιλήσει τελικά. Ορίστε εσεί τώρα δύο λεπτά. Julie Ward. Ναι, συγγνώμη, ε, δεν σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και για μένα προσωπικά, διότι εγώ στην πολιτική ε, μπήκα για να υπερασπιστώ την κοινωνική Ευρώπη, ιδιαίτερα για τους νέους. Τους νέους ε, στην εκπαίδευση, στην επίσημη αλλά και στην άτυπη και συναντώ συχνά νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικά ανήσυχοι για το μέλλον τους και έχουν την εντύπωση ότι τους κλέψαμε τις ευκαιρίες τους. Ε, εξετάζεται λοιπόν τι, θα, τι ενδέχεται να συμβεί στο μέλλον. Μιλάμε για τους νέους ανθρώπους ε, οι οποίοι ε, σχεδίαζαν να συμμετάσχουν σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και τώρα ε, νιώθουν ότι θα αποκλειστούν. Οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερα οι νέοι Βρετανοί που ήθελαν να έρθουν να σπουδάσουν στην Ευρώπη, ε, βλέπουν αυτή την ευκαιρία να χάνεται. Αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο του νέους που σπουδάζουν. Είναι και οι άτυπε μορφές μάθησης. Εγώ ε, έχω συνεργαστεί με αποκλεισμένους νέους ανθρώπους. Ε, υπάρχουν τεράστιε ευκαιρίε που ανοίχτηκαν για αυτού του ανθρώπου που συμμετείχαν σε διάφορα ειρηνευτικά ε, προγράμματα από πολλές χώρες, ε, άνθρωποι που δεν μιλούσαν καν την ίδια γλώσσα, αλλά ε, ζώντα μαζί για δύο εβδομάδες άλλαξε η ζωή τους. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς φοιτητές και μαθητές Υπάρχει ένα θέμα που σχετίζεται και με τη διαβίου μάθηση. Τώρα είπατε για το κόστος, είπατε για τα χρήματα, αλλά υπάρχει ένα ανθρώπινο κόστος. Και το ανθρώπινο κόστος ε, μας αφορά όλους. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία περίπτωση που, που αναφέρεται και στην εφημερίδα Guardian, ένα συνάδελφος, συντηρητικός βουλευτής, ε, φιλοευρωπαίος όμως, μου το έδειξε, είναι κάποιος από, τη δική του η λογική περιφέρεια στο Λάνκασερ, από την οποία προέρχομαι και εγώ, που ήταν καθηγητή σε ένα τοπικό ε, σχολείο το... και είπαν στο παιδί του πρέπει να φύγεις, να πας σπίτι σου και του πέταξαν, πέταξαν ένα τούβλο και σπάσαν το παράθυρο του σπιτιού του. Ε, δηλαδή η διαδικασία του Brexit αυξάνει και την ξενοφοβία, αυξάνει τον ρατσισμό. Και είναι κάτι το οποίο είναι συνεχές στη χώρα μου και είναι πραγματικά ντροπιαστικό και λυπηρό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Όλοι και όλες κατανοούμε τις ανησυχίες των νεαρών Βρετανών και Βρετανίδων σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Αλλά από την άλλη μεριά είναι βέβαια και οι επιπτώσεις της συμφωνίας, ε, της ε, άποψη της πλειοψηφίας που εκφράστηκε στο δημοψήφισμα. Υπάρχει καθαρή συμφωνία και των τριών θεσμικών οργάνων, δηλαδή Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής, ότι πρώτα θα συζητήσουμε την έξοδο και όταν πλέον θα έχει γίνει πλήρης η διαπραγμάτευση της εξόδου, της αποχώρησης και έχουν διευκρινιστεί τα ζητήματα του καθεστώτος που θα διέπει τους Ευρωπαίους πολίτες ε, στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και το ανάποδο, τότε θα συζητήσουμε πλέον πώς θα διαμορφωθούν οι μελλοντικές σχέσεις. Και αυτό βεβαίως πιάνει και όλα τα προγράμματά μας. Γι' αυτό και βρίσκω σωστό και σημαντικό να μην αναμειχθούν οι δύο αυτές συζητήσεις. Και βέβαια, από όσο θεωρώ, η Μεγάλη Βρετανία στο μέλλον κάποτε θα πρέπει και θα μπορεί να συμμετέχει στα προγράμματα. Βεβαίω με τις ανάλογες υποχρεώσεις και δικαιώματα και την δημοσιονομική συμμετοχή. Όμω, όπως είπα, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν ότι πρώτα συζητούμε το Brexit και όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το Brexit, τότε θα συζητήσουμε πλέον τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μεγάλη Βρετανία. Και νομίζω ότι και εμείς εδώ στην ομάδα εργασίας παρατήρηση του Brexit θα πρέπει να το τηρήσουμε. Παρόλοι, ξαναλέω, την πλήρη κατανόηση που έχω για την, ε, για τις ανησυχίες των νέων στην Μεγάλη Βρετανία. Όμως νομίζω ότι ο δρόμος που έχουν καθορίσει τα τρία θεσμικά όργανα είναι ο σωστός και μέσιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την ευγενική σας εισαγωγή. Είναι τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ. Τα θέματα πολιτισμού και παιδείας είναι ύψης της σημασίας και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης ε, μοιράζονται την κληρονομιά αυτή. Τώρα προχωρώντας, εγώ θυμάμαι προτού μπει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπήρχε υψηλό βαθμό συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την αλυσίδα. Υπήρχαν ανταλλαγέ σπουδαστών, φοιτητών κτλ και νομίζω ότι και σήμερα υπάρχει σημαντική συνεργασία και με πανεπιστήμια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν οφείλονται όλα αυτά τα προγράμματα ή στην Ένωση. Τώρα είναι σημαντικό, πιστεύω, στις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν μεταξύ ημών με ΙΤΑ και της Ενώσεως, ιδιαίτερα εσείς που είστε τα μέλη αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης, να βοηθήσετε ώστε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Νομίζω είμαι βέβαιος ότι και μετά θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ και επαφές μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδραμάτων των Βρετανικών και των Ευρωπαϊκών αλλά και των κυβερνήσεων. Θα έχουμε νέες πρωτοβουλίες, θα έχουμε νέες ευκαιρίες και είμαι σίγουρος ότι ο κοινό μας πολιτισμός θα πρέπει να βοηθήσει το κοινό αυτό πολιτιστικό πλαίσιο. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι η Πρόεδρος θα συμφωνεί μαζί μου ότι δεν θα συμμερίζονται όλοι οι συνάδελφοι όλα αυτά τα τρομακτικά που μας είπε η συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν δείχνουν κάτι τέτοιο τα μεγέθη. Μην εντυπωσιάζεστε λοιπόν από τέτοιου είδους σχόλια σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Ζαμπίνα Φαχάιμ δύο λεπτά. Νομίζω ότι η Επιτροπή Πολιτισμού δεν είναι ίσως η έδρα στην οποία θα πρέπει να διεξάγονται εσωτερικές συνομιλίες πολιτικού χαρακτήρα για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ έχουμε κάποιες επιπτώσεις, καταρχάς της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να δούμε ποια έχουν ήδη ολοκληρωθεί τον πραγματισμό του, ποια έχουν καταβληθεί κτλ. Όπως είπε και η Πρόεδρος, αυτό πρέπει να δούμε τώρα, είναι πώς θα διακρίνουμε με σαφή τρόπο μεταξύ των διαφόρων αυτών περιπτώσεων. Και δεν είναι ένα νησί που θα εξαφανιστεί η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένα νησί πολύ κοντινό μας. Και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, και θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και θα καταλήξει κάποια συμπεράσματα. Αλλά πριν από τα θέματα συνεργασίας ε, και που θα πρέπει να επιληθούν με λεπτομερή τρόπο, θα πρέπει να εστιαστούμε, να εντοπίσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, ποιες είναι οι συνέπειες, χωρίς ε, ευθύς εξ αρχής να λέμε, να, χαθούμε στη συζήτηση του τι θα γίνει στο μέλλον γενικός και ορίστε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στα προγράμματα της αρμοδιότητός μας, ώστε να ανασυντάξουμε και να αναπρογραμματίσουμε τις σχέσεις μας και τις επαφές μας και για το μέλλον. Αυτά ισχύουν και για τη δική μας Επιτροπή και για τα δικά μας θέματα αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα και για τα θέματα των μέσων ενημέρωσης. Όλα αυτά θα είναι δύσκολα, θα πρέπει να έχουμε σαφή όρια και πλαίσιο αυτής της εξόδου και θα πρέπει να έχουμε και μια σαφήνεια σχετικά με την ε, με το νομικό πλαίσιο και τις νομικές επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν εξ αρχής από την αρχή να ξεκινήσουμε να στήσουμε μια νέα συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα πρέπει και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο να δει με ποιο τρόπο θα τιμήσει τις δεσμεύσεις και τις υποχρέσεις που έχει αναλάβει. Στην πανεπιστημιακή έρευνα, για παράδειγμα, έχουν εγκριθεί συγκεκριμένα προγράμματα πολυετή, όπου έχουν ήδη δαπανηθεί κονδύλια και δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε τα τελευταία τρία έτη προγραμματισμού. Πρόεδρο. ευχαριστώ. Δεν έχω άλλου συγκεκριμένου. Ας... Α, Κριστίνα, άρα σε παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, ε, φίλοι πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπεις να μιλήσω. Ας λάβουμε υπόψη το εξή. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της Μπολόνια, δεν συμμετέχουν μόνο χώρες μέλη της Ένωσης, στην διαδικασία αυτή. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν και άλλες χώρες. Εδώ αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Με άλλα λόγια, εγώ συμφωνώ ότι πρώτα πρέπει να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες του χωρισμού, του διαζυγίου. Μια άλλη δυνατότητα είναι ένα είδος πρόγραμμα έρασμος συν, όπου πάλι δεν συμμετέχουν μονάχα σπουδαστές από χώρε μέλη. Ξαναλέω, πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες συνεργασίας, για παράδειγμα με πολιτιστικά ιδρύματα και ούτω καθεξής. Αυτά πρέπει να γίνουν. Βεβαίω και θα είναι δύσκολο να λάβει κανεί, να λάβει μια χώρα δηλαδή, χρήματα από τα προγράμματα αυτά, παρόλο που η συνεργασία συνεχίζεται. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένη ότι η monitoring group θα συνεχίσει να μας στηρεί ενήμερες και ενήμερους. Αλλά μήπως κύριε συνάδελφε θέλετε πάλι το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχά, ε, ναι, ε, σχετικά με την ερώτηση της συναδέλφου Κώστα για τους αυτοματισμούς που μας λείπουν σχετικά με την επιμήκυνση της παραμονής. Όμως δεν υπάρχει ακόμα αυτή η συμφωνία. Ίσως στο μέλλον να υπάρξει ένας κάποιος αυτοματισμός ή ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο να μην το δεχθεί αυτό. Εν πάση περιπτώσει σήμερα δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία και πρέπει επίσης να θυμόμαστε γιατί αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους χρηματοπιστωτικούς πρώτα απ' όλα, δημοσιονομικούς και επίσης επειδή δεν συμφωνούν στην βασική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας όχι του κεφαλαίου αλλά των πολιτών, των ανθρώπων. Επομένω, οι διαπραγματεύσει αυτέ υπό το πλαίσιο αυτό ή στο πλαίσιο αυτό θα είναι πολύ δύσκολε. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και εμείς, μεταξύ των οποίων και των νέων. Επίσης έχουμε το εκπαιδευτικό σύστημα την ανώτατη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι, το οποίο σύστημα είναι εκτιμητέο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτού του συστήματος επωφελούνται οι φοιτητέ, οι Βρετανοί, οι Ευρωπαίοι, αλλά και αυτοί που προέρχονται από άλλες χώρες και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό και να αντλήσουν τα ωφέλη που μπορούν να αντλήσουν. μέχρι τώρα είχαμε ένα σύστημα βάσει του οποίου ε, ε, ε, η χρηματοδότηση, οι υποτροφίες εδίδονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Στο μέλλον θα πρέπει να ξαναδούμε πώς θα δίδονται οι υποτροφίες αυτές, αλλά προς το παρόν στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης δεν έχει τεθεί κάτι τέτοιο. vielen, vielen herzlichen Dank. ευχαριστώ. Νομίζω ότι κύριε Στογεύσκη και εσείς και η Monitoring Group θα συνεχίσετε να μας τηρείτε ενήμερες. Το δε θέμα θα μας απασχολήσει ασφαλώς όλο τον επόμενο χρόνο και πιθανώς και το μεθεπόμενο. Τουλάχιστον το μισό. Έρχομαι στο θέμα υπαριθμών 5. Πρόκειται για την συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έχει υποβάλει σχετική πρόταση με νέα εκεί για την ανώτατη εκπαίδευση. Πρόταση επίσης για την υποστήριξη των χωρών μελών με την συλλογή δεδομένων σχετικά με τα επαγγέλματα που αναλαμβάνουν οι απόφητη για την στήριξη της εκπαίδευσης όλων των νέων και για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ώστε οι νέες και οι νέοι να αποκτούν τις γνώσεις που είναι αναγκαίες σε αυτές τις εποχές της παγκοσμιοποίησης αλλά και της ταχύτατης τεχνολογικής πρόοδου. Θεωρούμε αυτό το πακέτο προτάσεων της Κομισιόν πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό αποφασίσαμε να συντάξουμε έκθεση πρωτοβουλίας. Η διάσκεψη των Προέδρων θα εγγύψει το θέμα την επόμενη, στην επόμενη συνεδρία της, για την έγκριση δηλαδή της έκθεσης πρωτοβουλίας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Λίντς και τον κύριο Ντόριτς από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να μας αναπτύξουν το σημαντικό αυτό πακέτο ε, για το οποίο θα σας δώσουμε 15 με 20 λεπτά και αν θέλετε να λάβετε εσείς το λόγο πρώτα μοιράστε τον χρόνο μεταξύ σας όπως θέλετε αρκεί να μην, αρκεί να μην υπερβείτε τα 20 λεπτά Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκλησή σας αλλά και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την ε, ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής. Θα σας εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται και ε, για τις δύο ανακοινώσει πρόκειται για τον τομέα των σχολείων και των πανεπιστημίων, της ανωτάτης εκπαίδευσης δηλαδή και της μέσης εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να πούμε πρώτα ότι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε με τις δύο ανακοινώσει Πρόκειται για τις προτεραιότητες του Πρόεδρου Γιούνκερ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εκπαίδευση και ιδίω για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και για τον κεντρικό ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον, στη μόρφωση του μέλλον της Ευρώπης. Αυτή είναι η αφετηρία. Όλα τα θέματα, όπως απασχολησιμότητα, όπως καινοτομία, όπως η συμμετοχή στην ε, ζωή της κοινωνίας. Όλα αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ε, να εγκύψουμε πρώτα βαθιά στη μελέτη της εκπαίδευση. Και γι' αυτό προβαίνουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις που είναι και σαφώς στραμμένες προς το μέλλον γιατί περνούμε μέσα από μια κατάσταση οικονομικά πολύ δύσκολη όπου χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί και να υπερβούμε την κρίση και θέλουμε να, μια Ευρώπη που να προσφέρει περισσότερες ε, και πιο ίσες ευκαιρίες σε όλους ε, να φροντίσει την καινοτομία και ούτω καθεξής. Αυτό το δείξαμε και με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λέμε ότι χρειάζονται μαζικές επενδύσεις στη δημιουργία και στην διοχέτευση δεξιοτήτων και γνώσεων. Άλλωστε και με την ευκαιρία της 60ης επαιτίου των συνθήκων της Ρώμης είπαν και αρχή κρατών και κυβερνήσεων πώς φαντάζονται την Ευρώπη των 27 ως μια Ευρώπη όπου οι νέοι και οι νέες θα μπορούν να απολαμβάνουν την βέλτιστη, την άριστη δυνατή εκπαίδευση. Και κατάρτιση και επίσης και η έκθεση του Πασκάλ Λαμή για τις επενδύσεις στο μέλλον της Ευρώπης πάλι στον τομέα της εκπαίδευσης. Δηλαδή πρόκειται για όλα αυτά τα μεγάλα στρατηγικά θέματα που στρέφονται γύρω από το ίδιο θέμα, μέλλον και εκπαίδευση. Και αποτελούν τα θεμέλια για την κίνηση αυτή. Είναι σαφές ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε βέβαια όλοι ποια είναι η κατανομή, η των αρμοδιοτήτων καταρχήν αρμοδιότητα για την παιδεία είναι, ανήκει στις χώρες μέλη. Με μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και αρμοδιότητα, αλλά έχουμε και την ηθική υποχρέωση να προωθούμε την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, με ανταλλαγές καλών πρακτικών και με διαμεθοριακή αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων. Αυτή είναι και η οπτική, ε, ας πούμε, που διέπει τις ε, δύο ανακοινώσεις. Αφενός θεσπίζουν μεγάλους στόχους, από την άλλη μεριά τονίζουν ποιες είναι οι μεγάλες, οι τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει η σχολική εκπαίδευση και η συνάδελφός μου θα αναφερθεί στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Όταν μιλώ για τη σχολική εκπαίδευση και όταν εξετάζω τη σχολική εκπαίδευση, βλέπω από όλες τις μελέτες πόσο σημαντικό είναι να αρχίσει κανείς την προσπάθεια νωρίς την προσπάθεια της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό και για την επιτυχία της ίδιας της εκπαίδευσης, αλλά και για την επαγγελματική εξέλιξη των, ανθρώπων. ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση ε, στο, σε όλο το κοινό. Μάλιστα από την νεαρότατη ηλικία του παιδιού να μπουν οι βάσεις για να έχει το παιδί μετά και τη δυνατότητα να εποφεληθεί και από την διαβίου κατάρτιση και βεβαίως και από την περαιτέρω κατάρτιση των ε, ενηλίκων και θα έχει μια στέρεα βάση για να αντιμετωπίσει και τις ανάγκες του επαγγέλματος αργότερα. Δεύτερο, η εκπαίδευση είναι σημαντικός τομέας, όχι βέβαια, βέβαια μόνο για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές, είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα και τις οικογένειες. Επίσης, και όλες τις οργανώσεις, ε, τις κοινότητες, ε, δήμους και ούτω καθεξής. Πρέπει να δούμε λοιπόν πρώτα πια να κάνουμε μια καταγραφή της κατάστασης στην Ευρώπη. Και διαπιστώνει κανείς τον το πράξει αυτό ότι όντως υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ασφαλώς, αν κάνει κανείς μια σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, διαπιστώνει ότι η Ευρώπη υπαρέχει σε κάποιου τομεί, αλλού όμω αντιμετωπίζει σοβαρότατε προκλήσει. Αυτέ τι τονίζουμε στην ε, ανακοίνωσή μα ω εισαγωγή και οι τρει πιο σημαντικέ προκλήσει τι οποίε έχουμε συνοψίσει είναι ότι αφενός βλέπουμε δυστυχώ ότι το επίπεδο των ε, εκπαιδευτικών συστημάτων σε ό,τι αφορά την προώθηση των ικανοτήτων και των μαθητών αλλά και των ενηλίκων βλέπουμε ότι χρειάζεται βελτίωση, για να το πω απλά και καθαρά. Και ο τελευταίος γύρος πίσα, η πίζα, είδαμε ότι δεν έδωσε διόλου ενθαρρυντικές ειδήσει. Βλέπουμε σταθερότητα μέχρι πτώση και μάλιστα και απογοητευτικά αποτελέσματα για πολλές χώρες και στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Βλέπουμε ορισμένες χώρες μέλη οι οποίες τα πάνε πάρα πολύ καλά, βλέπουμε άλλες οι οποίες υστερούν πολύ. Τα αποτελέσματα λοιπόν της μελέτης PISA πραγματικά δεν είναι αυτά που θα θέλαμε να βλέπουμε από την Ευρώπη. Δεύτερο τομέα είναι η ισότητα των ευκαιριών. Εδώ εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι η εκπαίδευση και όπως είπα και μέσα από την μελέτη ή τις μελέτες PISA πολύ συχνά η εκπαίδευση απηχεί ή αντανακλά και τις, και τις κοινωνικές διαστρωματώσεις. Το τρίτο θέμα είναι η ψηφιοποίηση και η ταχύτατη ανάπτυξη τεχνολογίας. Επομένως, δεξιότητες, ισότητα ευκαιριών, ψηφιοποίηση. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα θέματα. Τι μπορεί να κάνει κανείς τώρα για να αντιμετωπίσει προκλήσεις αυτές. Εντοπίζουμε τα επίπεδα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, όπου έχουμε καλά παραδείγματα από ορισμένε χώρες μέλη, αφενός δηλαδή για παράδειγμα βάζουμε το ερώτημα πώς μπορούμε να προσφέρουμε στα σχολεία τις συνθήκες ώστε να λειτουργήσουν σωστά, να έχουν υπαρκείς πόρους, να συνεργαστούν και με εξωτερικούς φορείς, δεύτερο εκπαιδευτικό προσωπικό, πρέπει να ρίξουμε βάρος εκεί, δηλαδή χρειάζονται νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι ορισμένες φορές, υπάρχουν χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την περαιτέρω κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το ίδιο με τα μισθολογικά του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το τρίτο, που θέτουμε, το τρίτο ζήτημα που θέτουμε δηλαδή είναι ζητήματα governance, ζητήματα οργάνωσης, διοικητικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν είναι πάλι τα θέματα για τα οποία επιθυμούμε να συνεργαστούμε και με τι μέλη αλλά και με ομάδε συμφερόντων για να αναπτύξουμε κοινέ πολιτικέ και προτείνουμε στην βάση αυτών των τριών προκλήσεων και των τριών αυτών θεμάτων έναν αριθμό επιμέρου δράσεων, τι οποίε δεν θα αναπτύξω όλε τώρα με λεπτομέρεια, θα πω λίγα παραδείγματα μόνο. Για τον τομέα τη σχολική εκπαίδευση, για παράδειγμα, για μα είναι πολύ σημαντικό η κινητικότητα στην σχολική εκπαίδευση να μπορεί να συνεχιστεί και να ενταθεί. Μεγαλύτερη και καλύτερη κινητικότητα και μεταξύ σχολείων και διασύνδεση σχολείων, ηλεκτρονική δημοποίηση δηλαδή, και να συνεχίσουμε στην προσπάθεια αυτή. Έχουμε αναπτύξει και ένα tool, ένα μηχανισμό που θα τον συζητήσουμε, θα τον, θα τον ε, τεστάρουμε μάλλον το φινόπορο. Επιτρέπει να δούμε πόσο έχει προχωρήσει το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην προπαρασκευή του για την ε, ψηφιακή εξέλιξη σε ό,τι αφορά το, διδακτικό προσωπικό, δασκάλους, δηλαδή θέλουμε να συνομιλήσουμε με τις χώρες μέλη και με τους κοινωνικούς εταίρους, ιδίω για την εξέλιξη των σταδιοδρομιών των δασκάλων, πώς μπορεί δηλαδή το επάγγελμα να γίνει πιο ελκυστικό. Ποια μπορεί να είναι η περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη των δασκάλων και ε, των διδασκαλισών και βεβαίως διευθυντών σχολείων κλπ. Γίνονται πολλά πράγματα. Εκεί θέλουμε για τις χώρες εκείνες μέλη που ενδιαφέρονται, καθώς και για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται, να τους προσφέρουν μια πλατφόρμα ευρωπαϊκού διαλόγου. Τρίτο, για την governance, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή σκεπτόμαστε μαζί, σε συνεργασία με χώρες μέλη και για τις χώρες μέλη που το επιθυμούν, να τις ενισχύσουμε σε μια προσπάθεια εθνικής μεταρρύθμισης ώστε να προσλάβουν, να υιοθετήσουν καλές πρακτικές που γνωρίζουν από άλλες χώρες. Και σε συνεργασία και με τον ΟΟΣΑ. Ε, Εάν μια χώρα μέλος αποφασίσει για παράδειγμα ότι θέλει να εισαγάγει ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης των σχολείων του, να μπορέσει να κοιτάξει τι κάνουν άλλες χώρες μέλη στον τομέα αυτό. Αυτά με λίγα, πολύ λίγα λόγια για τον ε, τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και αν με επιτρέπετε να δώσω το μικρόφωνο στη συναδελφή μου, στη συναδελφό μου. Ευχαριστώ τώρα για ανώτερη εκπαίδευση. Θα περάσω στα αγγλικά αν δεν έχετε αντίρρηση. Η τελευταία μεγάλη πολιτική μας για τον τομέα αυτόν αφορά, ξεκίνησε το 2011, κάπως, δεν είναι και τόσο μακριά, μάλλον βοήθησε ε, τα κράτη-μέλη να επικεντρωθούν, να εστιάσουν ε, στους τομείς προτεραιότητας ε, όπου άλλους διαρρέθηκαν και τα χρήματα του Erasmus Plus, όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και λόγω της τεχνολογίας αλλάζει ο τρόπος εργασίας και ο χώρος εργασίας στον οποίο βρίσκονται οι απόφοιτοι της ε, ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και η οργάνωση. Υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός από ποτέ σε ό,τι αφορά τους αποφύτους αυτούς που ψάχνουν θέσεις εργασίας από την Κίνα, την Ινδία, από παντού στον κόσμο. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να φανεί, πιο καινοτόμα από ποτέ. Εμείς θεωρούμε ότι οι θεσμοί της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όλο και πιο σημαντικό ρόλο στον τομέα της δημοκρατικής ζωής εκεί όπου υπάρχει ε, υπάρχουν όλο και περισσότερες προκλήσεις πρέπει η εκπαίδευση, η επιστήμη να αποκαταθεί εμπιστοσύνη προς αυτές ε, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη και τα ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει αυτέ. Εμεί σεβόμαστε βεβαίω την αρχή τη επικουρικότητα σε ό,τι αφορά τον τομέα τη εκπαίδευση. Η ατζέντα μας λοιπόν έχει τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μελλοντικών προσόντων που δεν θα συνάδουν με τις ανάγκες σε προσόντα. Ε, να έχουμε συστήματα ανώτης εκπαίδευσης που να είναι συμπεριληπτικά, διότι ε, συνήθως η ε, μεσαία τάξη και πάνω φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση και τα παιδιά του ε, πιο κάτω δεν φτάνουν και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επίση πρέπει να είναι πιο συνδεδεμένοι με τον πραγματικό κόσμο. Η ανώτατη εκπαίδευση, με την κοινωνία των υπάρχουν και κάποιε δεξιότητε κοινωνικέ που πρέπει να αναπτύξουν οι φοιτητέ. Θέλουμε η ανώτατη εκπαίδευση να συνεισφέρει πιο αποτελεσματικά και στην καινοτομία, για στι περιφέρειε όπου βρίσκονται αυτά τα ιδρύματα. Επίση, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα αυτά θα είναι και αποτελεσματικά και λειτουργικά έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι πόροι, να διατίθενται οι πόροι με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε λοιπόν και εμεί μια σειρά δράσει για να επιτευχθούν αυτοί οι τέσσερι στόχοι. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε όλου του στόχου, σε όλε τι δράσει προφανώ, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μια δράση που για μα είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι η υποστήριξη τη ε, εκπαίδευση, τη μάθηση και τη. Ε, ε Θέλουμε δηλαδή το προσωπικό, το εκπαιδευτικό να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύεται το ίδιο. Ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Erasmus Plus ακόμα περαιτέρω έτσι ώστε το ε, καθηγητικό προσωπικό να μπορεί ε, να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτό έχει να κάνει και με πρωτοβουλίες για καινοτόμα βιογραφικά που θα βοηθούν ε, μάλλον καινοτόμες, ε, καινοτόμα μαθήματα σε, στα πανεπιστήμια που να δίνει πρόσβαση και σε ανθρώπους που εργάζονται, σε ανθρώπους που ακολουθούν εναλλακτικέ οδούς μάθησης, ε, μεγαλύτερη κινητικότητα, όλα αυτά θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα. Επίσης θα εξετάσουμε τα συστήματα ανώτατη εκπαίδευσης στο σύνολό τους, περιλαμβάνοντας και το πώς κατανείμονται οι πόροι τα θεσμικά όργανα και μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων, πώς δηλαδή η, ε, στηρίζεται η, η καθηγητική δραστηριότητα σε σχέση και με την έρευνα θα πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές ό,τι φορά το τι φοιτεί ο καθένας ε, και θα πρέπει να καλύψουμε τις ελλείψεις. Ε, υπάρχουν κάποιοι τομείς κλειδιά, αλλά ε, αναγνωρίζουμε το έγγραφό μας ότι πρέπει να προσαρμοστούμε, να πρέπει να έχουμε μάλλον φοιτητέ που να μπορούν να προσαρμόζονται σε μια κοινωνία που αλλάζει. Και αυτό απαιτεί μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερα προσόντα τα οποία είναι διατομιακά και μεγαλύτερε δυνατότητε προσαρμογή σε ε, μια ζήτηση η οποία αλλάζει. Ε, πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε και την τέχνη σε αυτές τις βασικές δεξιότητες Τέλος, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ε, προσόντα στις δεξιότητες που ε, αποκτούν οι μαθητές και πώς θα μετρώνται αυτές οι, οι δεξιότητες. Να υπάρχει μια παρακολούθηση δηλαδή για να μπορούμε να προσμετρήσουμε και την ποσότητα και την ποιότητα και τι είναι στη θέση να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν ε, φεύγουν από την άλλη εκπαίδευση. Αυτά σκοπεύουμε λοιπόν για την άλλη εκπαίδευση να υλοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, κάτι άλλο. Νομίζω ότι εμπίπτει στην ευρύτερη προσέγγιση αυτό. Δεν πρέπει να το δούμε αυτά απομονωμένα. Νομίζω ότι εντάσσονται στην ευρύτερη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη των νέων ανθρώπων. Αναμένουμε λοιπόν με ανεπιμονησία την συνεργασία μα μαζί σα για την εφαρμογή τη και περιμένουμε και τι ιδέε σα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει η για αυτήν την συνολική εικόνα που μας ε, διαβιβάσατε, που μας περιγράψατε και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Λιμπάτσκα και θα ακούσουμε και τους ε, σκιώδεις ακολούθως και τους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Κύριε κυρία Λιμπάτσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε, τώρα σε δύο-τρία λεπτά θα δυσκολευτώ λιγάκι, αλλά θα προσπαθήσω. Τώρα ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ για την ενίσχυση που εκφράσατε την υποστήριξη ε, στα εκπαιδευτικά συστήματα. Είμαι σύμφωνη με εσάς ότι για να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ε, χρειαζόμαστε, πρέπει να στηριχτούμε πάνω στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και νομίζω ότι σχετικά με αυτό είναι υπεύθυνοι και οι Υπουργοί Οικονομικών, αυτοί που είναι αρμόδιοι για τα δημοσιονομικά. Γιατί συμφωνούμε όλοι, όλοι τοποθετούμαστε με τον ίδιο τρόπο για τις βασικές αρχές, αλλά μετά όταν πάμε ε, στα συγκεκριμένα ζητήματα στο Erasmus βλέπουμε ότι δεν προχωρούμε, δεν επιτυγχάνεται συμφωνία, είμαστε ελληματικοί. Στην Επιτροπή μας εμείς ε, θέλουμε ακριβώς να λάβουμε υπόψη μας ε, τις θέσεις που εκφράσατε και έχουμε ε, προτείνει τέσσερις δέσμες προκειμένου να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Μία πρώτη δέσμη είναι τα διάφορα πεδία της κατάρτισης στο οποίο συμβάλλουν τα δημοσιονομικά, η οικονομία, η ανάπτυξη, όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή εκτός του εκπαιδευτικού και συστήματος, συστήματος κατάρτισης. Τώρα δεύτερη δέσμη για τα διάφορα συστήματα στην Ευρώπη. Μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων πρέπει να βρούμε την επαφή μεταξύ των συστημάτων αυτών, όπως και την εγκατάλειψη των σπουδών. και έχουμε διάφορες πηγές ενημέρωσης Η τρίτη δέσμη είναι εκείνη των ε, διδασκόντων, των ε, δοκίμων ε, καθηγητών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα ρόλο τελείως διαφορετικό δεν είναι η μοναδική πηγή ενημέρωσης όπως ήταν στο παρελθόν ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να είναι απλώς καταρτισμένοι και ενημερωμένοι θα πρέπει να έχουν και δεξιότητες που είναι πλέον απολύτως απαραίτητες όπως οι ψηφιακές αυτό έχει άμεση σχέση με, την, με το ρόλο των καθηγητών. Οι δόκιμοι διδάκτορες ή καθηγητές ή διδάσκοντες πρέπει να διαμαντήσουν το πιο δυναμικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. για το μέλλον θα πρέπει να έχουμε διδακτικό προσωπικό που να αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η οικονομία, η κοινωνία, ο κόσμος και να μπορούν και να τη διαμορφώνουν. Οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες όποια και να είναι η δεσμευτικότητα ή η υποχρεωτικότητα του συστήματος. Εμείς έχουμε προβλέψει μια σειρά από συναντήσεις μεταξύ των ενώσεων των καθηγητών και των σπουδαστών. Θα είναι όμως και σημαντικό στη συνεδριά της Επιτροπής να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους και ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να στηριχτούμε και στη δική σας εισφορά. Σας ευχαριστώ Κριστίνα, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Μπότσκορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα ελέγχθησαν ε, από τους συναδέλφους πριν από μένα. Υπάρχουν ε, δύο σημαντικά. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε εμείς για τα θέματα της αρμοδιότητός μας, αλλά υπάρχει και η εξής ιδιαιτερότητα. χρειαζόμαστε μια ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Υπάρχουν χώρες με πετυχημένα και δυναμικά συστήματα που μπορούν να δώσουν το παράδειγμα για τις χώρες που αντιμετωπίζουν καθυστέρηση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι όταν αφιερωθούν τα, τα απαραίτητα κονδύλια έχουμε αποτελέσματα. Απουσία πόρων, απουσία κονδυλίων δεν μπορούμε να έχουμε επαρκή αποτελέσματα. Και έχουμε και εκνευρισμό και ανησυχία των διδασκόντων. υπάρχει τρόπος να βελτιώσουμε τη συνολική ποιότητα του, του εκπαιδευτικού συστήματος. Και συμφωνώ με τους παραλύσαντες ότι πρέπει να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε το συνολικό επίπεδο το σχολικό. Και με αυτό δεν εννοούμε να ασκήσουμε πίεση στους μαθητές, εννοούμε να έχουμε ιδρύματα, σχολεία, που θα δίνουν κίνητρα, που θα δίνουν τις απαραίτητες βάσεις στα παιδιά. Να τους δίνουν δηλαδή τις, τα θεμέλια ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, τις γλωσσικές, ε, τις ψηφιακές και όλες τις υπόλοιπε. Είναι οι βασικές γνώσεις που θα πρέπει να ε, έχουν τα παιδιά για το υπόλοιπο της ζωής τους και για την καθημερινή τους ε, ζωή και για τις ε, ευθύνες τους ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. με έναν τρόπο ώστε να κεντρίζεται και η περιέργεια, αν θέλετε, η απολύτως φυσική περιέργεια του παιδιού, για να πτήσει τις δυνατότητες του. Επίση είναι σημαντικό η σταδιοδρομία των διδασκόντων να είναι ελκυστική για του νέου, Όχι ώστε να καταλήγουν και οι άνθρωποι που, που απλώς δεν μπορούν να βρουν καμιά άλλη δουλειά, αλλά να έχουμε πραγματικά κίνητρα. Να είναι ελκυστική η σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ. Κυρία. Δύο λεπτά σας παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου ομιλεί Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή γιατί είναι ένα από τα θέματα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ λέω ότι εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ε, παρά τις επικρίσεις λοιπόν που ακούμε συνεχώς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ τα πράγματα είναι αντίστροφα. Έχουμε και την κυρία Κώστα και τον άλλο Ιταλό συνάδελφο εδώ τους οποίους επικαλούμε, αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, χώρα που ίδρυσε και αυτή την Ευρώπη. Ε, ε, βλέπουμε φαινόμενα λοιπόν στη χώρα μας που είναι εξαιρετικά ανισχυτικά. Το Σύνταγμα μας έχει ένα πολύ ιδιαίτερο άρθρο που λέει ότι η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από το κράτος αλλά ή και από την κοινότητα. Αλλά σχετικά με τη χρηματοδότηση δεν είναι σαφές το άρθρο του συντάγματος. Το πιο ενισχυτικό βέβαια δεν είναι αυτό. Είναι ότι αρχίζουν να εμφανίζονται σχολεία της υποχρεωτικής παιδείας που αρχίζει να σχηματίζεται ένα σκηνικό βάση του οποίου κάποιοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα σχολεία αυτά τις οικονομικές και άλλοι απλά δεν τις έχουν. Αρχίζει και χωρίζεται η χώρα στα δύο. Και νομίζω ότι αυτό που ανισχύει το σύνολο της Ευρώπης, ότι αυτά τα βλέπουμε όχι μόνο στις σχολείες, όχι μόνο στην εκπαίδευση δηλαδή, αλλά και στα θέματα κατοικίας. Αρχίζουμε και βλέπουμε κτίρια με εξι μέτρα τείχο γύρω-γύρω, ώστε να προστατεύσουν το κάλος ή την κομψότητα της συγκεκριμένης κατοικίας του συγκεκριμένου κοντομίνιου. Αυτά μας οδηγούν σε πολύ ανησυχητικές καταστάσεις. Ακούμε ότι δεν μπορεί κανείς να είναι διδάσκον όταν δεν γνωρίζει ένα επάγγελμα του αρχιτέκτονα, του μαθηματικού, του οποιοδήποτε άλλου. Εγώ πιστεύω ότι η επένδυση στην ποιότητα του διδάσκοντα, ο ενθουσιασμός του για να διαβιβάσει τη φλόγα αυτή στα παιδιά, γιατί μια χώρα είναι τόσο δυναμική ή μια κοινωνία είναι τόσο δυναμική όσο πιο ψηλά τοποθετεί στην ιεραρχία της ε, την παιδεία. Και έχουμε και ένα θέμα το οποίο έχουμε παραμερίσει μερικές φορές, ε, το θέμα της οικογένειας. Έχουμε το σύστημα της Δανίας που την λαμβάνει πολύ σημαντικά υπόψη της και το δικό μας σύστημα που την λαμβάνει πολύ λίγο υπόψη της, την οικογένεια. Αλλά χρειαζόμαστε όλα αυτά τα στοιχεία για να φτάσουμε ίσως σε αυτό το όραμα που πριν από 70 χρόνια κάποιοι είχαν για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κυρία Σάντοβα. Děkuji za vysvětlení, za e, předložení tohoto tématu. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι βέβαιος αν μιλάμε τελικά για το έγγραφο της Κομισιόν ως πολιτικό έγγραφο ή αν μιλάμε για τη μελέτη. σχετικά με την αόρατη εκπαίδευση. Μιλάμε σε διάφορα επίπεδα και δεν είναι σαφές για μένα. Εγώ δεν έχω την ανακοίνωση μπροστά μου. Για ποιο έγγραφο τελικά μιλάμε. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Θα ήθελα να ξέρω επίσης πώς συνδέεται αυτή η ανακοίνωση με τη νέα ατζέντα για τις δεξιότητες και τα προσόντα, που είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο κατά τη γνώμη μου. Δεν βλέπω όμως πώς συνδέεται αυτό. Η ατζέντα με τις, ε, για τις νέες δεξιότητες αναφέρεται σε 7 νέα μέσα. Κάποια αφορούν και τον εξοχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Αλλά δεν αναφερθήκατε σχετικά. Δεν είπατε δηλαδή θα χρησιμοποιήσετε στοιχεία ή ε, μέσα εργαλεία από την ατζέντα σχετικά με τις νέες δεξιότητες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πιο σφαιρική. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε συνέχεια νέε ανακοινώσει και να μην ξέρουμε πώ συνδέονται μεταξύ του. πιστεύουμε ότι η ατζέντα είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσο εφαρμόζεται τελικά αυτά τα συμπεράσματα και αυτά οι συστάσει που προκύπτουν. Θα ήταν πραγματικά καλό να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Τρεις ακόμα έχουν στήσει το λόγο και στη συνέχεια θα κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών. Julie Watt, για δύο λεπτά, παρακαλώ. Julie Ward. Δεν θα χρειαστώ δύο λεπτά νομίζω. Ήθελα απλώς να πω ότι χάρηκα που άκουσα ε, ότι ε, η έννοια του STEAM προχωράει, διότι για πολύ καιρό το STEM έχει αφήσει εκτός τα ζητήματα τα καλλιτεχνικά, την τέχνη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούστηκε αυτό έτσι με φυσικότητα κιόλας διότι εφόσον το έχει κατά νου αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έχουν κατά νου οι πολιτικοί θύνοντες, οι ερευνητέ, η ακαδημαϊκή κοινότητα, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα βεβαίω οι προκλήσεις παραμένουν. Θα πρέπει κάπως αυτό να φτάσει και στα αυτιά των εργοδοτών. Πέρα δηλαδή από την εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όσοι ε, εργάζονται στη συνέχεια στον χώρο εργασίας θα καταλάβουν τη σημασία του STEAM είναι κάτι σημαντικό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάμιτ τώρα έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή προηγουμένως και την, το καλωσόρισμα ουσιαστικά. Ήμουν πρώην Υπουργό Πολιτισμού και έχω παρακολουθήσει τα ζητήματα αυτά σε εθνικό επίπεδο και τώρα βεβαίως με μεγάλο ενθουσιασμό αναμένω να συνεισφέρω και εγώ στη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μα. ορίζω την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, διότι όταν συζητάμε για την ανάγκη εξχρονισμού τη εκπαίδευση, αυτό μου σημαίνει, ε, μου θυμίζει μάλλον, ότι συχνά ε, η εκπαίδευση είναι ένα κλειδί για πολλές πόρτες, για την καινοτομία, την ανάπτυξη ζωής, την, την, ανάπτυξη, την οικονομική μάλλον, την ε, κοινωνική ζωή. Ε, μίλησαμε για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, των καθηγητών. Και σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, και τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να αναφερθώ στο πόσο εγώ καλωσορίζω τις προσπάθειες που γίνονται από την, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εκπαίδευσης στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των ακαδημαϊκών. Χρειάζεται μεγαλύτερη επικοινωνία και χρειάζεται εκπαίδευση για να μπορεί να λάβει χώρα αυτή η επικοινωνία. Η σημασία των καθηγητών πρέπει να τονιστεί και να συνδυαστεί με το να θεωρηθούν οι καθηγητές εμπλεκόμενοι φορείς. Πρέπει ήδη να οικειοποιηθούν την όλη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο και περισσότερο διάλογο με τους ε, καθηγητές. Ό,τι αφορά τώρα τους φοιτητές, τους μαθητές, θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικά τα προγράμματα, να είναι πιο ενδιαφέροντα, να είναι πιο ε, διασκεδαστικά, αν θέλετε. Νομίζω ότι όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν και δημιουργεί πολλές προκλήσεις για μας για το μέλλον. Ευχαριστώ, κυρία Ιμπάνιεθ. Ε, κυρία Κώστα, συγγνώμη. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Κομισιόν, έστω και με καθυστέρηση, ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την στρατηγική Ευρώπη 2020, ε, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση. Είναι κάτι που το είχαμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε το σύνολο του πλαισίου, τις διάφορες προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και την επικουρικότητα. Εδώ υπάρχει και το θέμα της βασικής εκπαίδευσης, των σχολείων δηλαδή, ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε εμείς ένα νέο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό έχει επιπτώσεις και στην αποσχολησιμότητα των φοιτητών, των απόφοιτων. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα, ένα μέσο παρακολούθησης. Στα πλαίσια αυτών των δύο ανακοινώσεων αναφερθήκατε σε κάποια κεντρικά σημεία από την οποία θα πρέπει να εργαστούμε. Είναι σωστά όλα αυτά. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ε, ο κύριος Αλιμπάσκα. Ε, είναι τρεις εκθέσεις, αλλά τα ζητήματα είναι οριζόντια σε όλες τις ανακοινώσεις, σε όλες τις εκθέσεις. Και κάτι ακόμα. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε για εξχρονισμό να συμπεριληφθούν τρία παραδείγματα. Η συμπερίληψη, η συμπεριληπτικότητα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτό, διότι οι ανισότητες είναι ένα πρόβλημα στο οποίο δεν δίνει απάντηση το σχολείο. Και οι διαφορές σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες μεγαλώνει ακόμα περισσότερο μετά την ε, πανεπιστημιακή ζωή και καθώς προχωράμε προς την επαγγελματική ζωή. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί το θέμα της διακυβέρνησης. Να λοιπόν τρία ζητήματα πολύ σημαντικά τα οποία θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα εμάς τους ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους λεγόμενους βέβαια για το ζήτημα αυτό. Δύο λεπτά κύριε Μοργάνο. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω δύο-τρία σχόλια. Ναι, χρειάζεται ένα πλαίσιο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε μία εξίσωση, μία εξισορρόπηση. Η θα έχουμε μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των δεξιοτήτων. Πρέπει να είναι σαφή τα κείμενά μας. Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει μέχρι ένα σημείο. Πρέπει εμείς όμως τα προγράμματα να τα Πρέπει τα διάφορα μαθήματα να τα φέρουμε πιο κοντά. Έτσι ώστε να έχουμε ένα πραγματικό χώρο εκπαίδευση στην Ευρώπη. Επίσης η διεθνοποίηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε και εδώ να συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας και κάτι το οποίο αναφέρθηκε ήδη πολλάκις, πώς θα δώσουμε κίνητρα τους α, ε, ανθρώπους να πάνε προς τον, χώρο της εκπαίδευσης, προς τον χώρο δηλαδή των εκπαιδευτικών, πώς κάποιος θα θελήσει να γίνει εκπαιδευτικός. Έχει σημασία πώς προσλαμβάνεται ο καθηγητής στην κοινωνία μας σήμερα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το θέμα της συμπερίληψης επίσης είναι σημαντικό, αλλά και αυτό αφορά την βελτίωση του επίπεδου εκπαίδευση. Είναι σαν τους λίγους ε, τρόπους που έχουμε έτσι ώστε οι πιο μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες να μπορέσουν να ανέλθουν κοινωνικά η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω δύο φράσεις κι εγώ. Για να είμαι ειλικρινής, παρόλη την επικουρικότητα δεν θα μπορέσει βεβαίω ποτέ να υπάρξει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα εκπαίδευση, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αλλά τι άραγε εμποδίζει τι χώρε μέλη να συνεννοηθούν και να συμφωνήσουν πάνω σε κάποιου κοινού ευρωπαϊκού στόχου εκπαίδευση. Και μπορεί να δει κανεί αν μπορούν να επιτευχθούν. Έχω κουραστεί λίγο να ακούω ξανά και ξανά από τους εθνικούς ε, διάφορους πολιτικούς των, των χωρών μελών δηλαδή πόσο σημαντική είναι η παιδεία, η εκπαίδευση κλπ. Και μετά να μην εξοπλίζουν την παιδεία με τους αναγκαίους πόρους ώστε τελικά να γίνει χρήσιμη για όλους. Έχω κουραστεί να τα πω αυτά τα πράγματα. Ίσως μπορούμε να περιλάβουμε στην έκθεσή μας και μια αξίωση που να απευθυνθεί στι χώρες μέλη και να πούμε δηλαδή ότι ένα ποσοστό του προϋπολογισμού της κάθε χώρας θα πρέπει να κατευθύνεται στην παιδεία. Τώρα βέβαια μένει το δικό μας πρόβλημα, το γερμανικό που είμαστε όπως είπα, ομοσπονδιακή χώρα, να δούμε πώς θα το πετύχουμε εμείς αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο. Αλλά να δοθεί ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν μιλούμε μονάχα, δεν λέμε μονάχα λόγια για επενδύσεις στην παιδεία. Αλλά να κάνουμε μια προσπάθεια να μπουν στόχοι και να τηρηθούν οι στόχοι αυτοί. Να δώσω πάλι το λόγο στην ε, κυρία Λίντσου και στον κύριο Τόιτς. Ένα λεπτό η Κριστίνα. Αγαπητή Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επειδή οι χώρες μέλη έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δυσκολότερα θέματα και συμφωνήσανε μάλιστα να συγχρηματοδοτήσουν και στρατιωτικό σύμφωνο. Γιατί όχι λοιπόν ένα σύμφωνο για την παιδεία. Ο κύριος Στόιτς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, αφού ευχαριστήσω πρώτα για τις υποδείξεις και χαίρομαι πολύ για την ε, διαγραφόμενη μελλοντική συνεργασία. Άκουσα για την ε, διάσκεψη που ε, οργανώνεται και πολύ ευχαριστώ να συνεργαστούμε κι εμείς. Θα επαναλάβω αυτό που είναι σημαντικό για μας, από, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, να ακούσουμε και από σας και από το Συμβούλιο αν η ανάλυση που υποβάλλουμε, κατά τη γνώμη σας, κινείται προς την ορθή πολιτική κατεύθυνση. Μιλούμε δηλαδή για την παιδεία μέσα στην συνολικότερη, ευρύτερη εικόνα με τις διάφορες διακλαδώσεις στον κοινωνικό τομέα, στην καινοτομία, στην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι η συμβολή της παιδείας σε όλα αυτά να καταστεί σαφές το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η προσπάθεια αυτή. Μιλήσαμε και για κάποιε προκλήσεις. Εσείς προσθέσατε και άλλε προκλήσεις. Η συμπερίληψη δηλαδή, ο μη αποκλεισμό όλων στην ε, εκπαίδευση, ε, τα θέματα των δασκάλων. Ερώτηση λοιπόν που απευθύνω προς εσάς. Θεωρείτε ότι έχουμε ε, εντοπίσει και περιγράψει σωστά τις προκλήσεις. Εξάλλου, έχουμε την πρόθεση σε ορισμένους τομείς όπου έως τώρα έχουμε συνεργαστεί με συναδέλφους μας των εθνικών κυβερνήσεων και εκπροσώπους διαφόρων οργανώσεων, ομοσπονδιών κλπ. Και σε ό,τι αφορά δηλαδή για παράδειγμα τις σταδιοδρομίες. Όλα αυτά που γράφουμε στις ανακοινώσεις μας δεν έρχονται από το μηδέν, είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο και με ειδικού από τις χώρες μέλη. Ελπίζω λοιπόν ότι οι προτεραιότητε όπω τις καταγράφουμε σας βρίσκουν σύμφωνους και αναμένω βεβαίω με μεγάλο ενδιαφέρον και το feedback που θα μπορέσετε να μας δώσετε. Η κυρία Λίντς. Τι άλλο να προσθέσω. ασφαλώ θα συνεργαστούμε στενότερα για τις λεπτομέρειες καθώς θα λαμβάνει πιο πλήρη μορφή η έκθεση. Συμφωνούμε με τι γενικέ γραμμέ που σας ενδιαφέρουν και εσάς. Είναι πολύ κοντά και στις δικές μας απόψεις Εάν χρειάζονται διευκρινήσεις για συγκεκριμένες δράσεις που προτιθέμεθα να προωθήσουμε, πολύ ευχαριστώ λοιπόν να δώσουμε σχετικές διευκρινήσεις, να διευκρινίσω ωστόσο, μιλούμε εδώ για την ανακοίνωση, όπως είπε όμως και ο Μιχαήλ, δεν έρχεται από το πουθενά. Προέρχεται από την εργασία που έχει προηγηθεί και από την ατζέντα για τις δεξιότητες. Ξαναλέω λοιπόν, δεν έρχεται από το πουθενά. Υπάρχουν υποστηρικτικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται η ανακοίνωση. Αλλά βεβαίω εδώ μιλούμε καθαρά για το περιεχόμενο των ανακοινώσεων. Και πολύ ευχαρίστω συνεργαστούμε μαζί σα. Η πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Μου φάνηκε πολύ χρήσιμη η συζήτηση και ω βάση για τι περαιτέρω συζητήσει και ελπίζω πολύ η διάσκεψη των πρόεδρων πολιτικών ομάδων να εγκρίνει την έκθεση πρωτοβουλία στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας. Δεν βρίσκω βέβαια να υπάρχει κανένα επιχείρημα κατά. Αναμένω λοιπόν συνεργασία μαζί σας για τα θέματα αυτά που νομίζω ότι είναι σημαντικά για όλες τις χώρες μέλη και εάν θέλουμε ως Ένωση να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και ίσως να μπορέσουμε να σπρώξουμε και λίγο για τις χώρες μέλη προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, νομίζω ότι αν το πετύχουμε αυτό, εξυπηρετούμε όλους τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες. Ευχαριστώ λοιπόν για την σημερινή σας παρουσία και την ανάπτυξη των σκέψεών σας και αναμένω με ενδιαφέρον την περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία και με εσάς, Επιτροπή δηλαδή, αλλά και με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως Πρόκειται για την ενημέρωση σχετικά με τον τριμερή διάλογο, σχετικά με την οδηγία τη υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων, που γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Άρα θα παρακαλέσω όλες και όλου όσοι δεν είναι μέλη τη ε, Επιτροπή Πολιτισμού ή δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, εδώ εννοώ και όλε και όλου του συνεργάτε τη Επιτροπή και δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου.